Good morning, uh, dear colleagues. I Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Θα πρότεινα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Έχω και κάποιες παρατηρήσεις και ανακοινώσεις ε, και όσο τις κάνω ελπίζω να συνδεθούν και άλλοι συνάδελφοι. Καταρχήν, ε, το σημείο είναι της ημερήσεις διάταξη, έγκριση της ημερήσεις διάταξης, θα πρότεινα δύο αλλαγές. Η πρώτη αφορά την ψηφοφορία για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων στα πέντε προγράμματα του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ. Την ψηφοφορία αυτή θα την αναβάλουμε για την επόμενη μα συνεδρίαση της 4 η Ιουνίου του 2020. Δεύτερη τροποποίηση είναι ότι μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για τις τρεις γνωμοδοτήσεις για τα δάση, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις με το σημείο 14, τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα. Θα ακολουθήσει το σημείο 12 για τη νέα ε, βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη και τέλος θα συζητήσουμε το σημείο 13, την ανταλλαγή απόψεων δηλαδή με διάφορους ομιλητές για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σας ευχαριστώ. Σύντομες ανακοινώσεις συνήθως μεταδίδεται στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και έχουμε διερμηνία σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά και πολωνικά. Παρακαλώ λάβατε υπόψη ότι οι διερμηνείς ε, στηρίζονται στην καλή ποιότητα του ήχου και της εικόνας της συνδέσεις των συμμετεχόντων εξ προκειμένου να διαβιβάσουν και να μεταφράσουν στα το μήνυμά σας. Γι' αυτό ε, μιλάτε κατά το δυνατό τις γλώσσες που υπάρχουν διαθέσιμες σε φυσιολογικό ρυθμό, αργά, καθαρά, ευδιάκριτα και να μπορέσουν να κάνουν σωστά το έργο τους οι διερμηνείς, τους οποίους ευχαριστώ εκ των προτέρων για την εργόδη προσπάθειά τους. Περνάμε στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας της 28 Απριλίου του 2020. Εγκρίνονται και περνάμε στις ε, ψηφοφορίες. Θα ψηφίσουμε τρεις γνωμοδοτήσεις. Η πρώτη αφορά το νέο πλαίσιο, νομικό πλαίσιο για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψήλωσης ε, που, στην οποία συνέβαλε και η Ευρωπαϊκή Ένωση παγκοσμίω. Δεύτερο αφορά την ε, στρατηγική για τα δάση και τρίτη την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη. Ο κύριος Πεκάρινεν είναι από την ομάδα Renew ο συντάκτης των γνωμοδοτήσεων με πολλούς και οδησηγητές. Σήμερα θα κάνουμε την τελική ψηφοφορία για τις τρεις γνωμοδοτήσεις και πριν περάσουμε στην έναρξη της ψηφοφορίας θα πρέπει να εξακριβώσουμε την απαρτία. Χρειαζόμαστε ένα τέταρτο των παρόντων μελών, δηλαδή 20 μέλη για να συγκεντρώσουμε απαρτία. Και για να την επιβεβαιώσουμε, παρακαλώ, πατήστε το κουμπί Raise Hand για να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τουλάχιστον 20 παρόντες. Εγώ είμαι βέβαιος ότι έχουμε την απαρτία, αλλά θα πρέπει να το ελέγξουμε. Παρακαλώ, συνάδελφοι, πατήστε το κουμπί Raise Hand. President, we have the Έχουμε απαρτία, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Οπότε περνάμε στην ψηφοφορία. Γνωρίζετε τους κανόνες, να τους επαναλάβω εντάχει. Μόνο οι ευρωβουλευτέ, των οποίων τα ονόματα έχουν ανακοινωθεί εγκαίρω ε, στη γραμματεία από τι πολιτικέ ομάδε, δικαιούνται να ψηφίσουν. Μπορείτε είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα να, σημειώσετε το ψηφο... να συμπληρώσετε το ψηφοδέλτιο. Ε, εκτυπώστε το, συμπληρώστε το όνομά σα, υπογράψτε την ε, επίσημη δήλωση. Μπορείτε να το σκανάρετε, να το φωτογραφίσετε και ενδεχομένω να το υπογράψετε και ηλεκτρονικά. Ε, και στείλτε το στην ε, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας έχουμε δώσει. Και μάλιστα στείλτε το από την επίσημη διεύθυνση ε, ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να ληφθεί υπόψη ως έγκυρη ψήφος. Βλέπω και πολλούς συναδέλφους στην αίθουσα και χαίρομαι ιδιαίτερο που είναι στις Βρυξέλλες. Και εφόσον είναι στον κατάλογο που έστειλαν οι πολιτικές ομάδες, μπορούν να επιδώσουν απευθείας στη γραμματεία το ψηφοδέλτιό τους. Κυρίσω την έναρξη της ψηφοφορίας και θα λάβετε mail από τη γραμματεία για να σας ζητήσει να ψηφίσετε. Μέχρι τη 1.30 ώρα Βρυξελών είναι η προθεσμία για την υποβολή του ψηφοδελτίου. Μέχρι τότε θα πρέπει να το στείλετε για να ληφθεί υπόψη. Και φυσικά η γραμματεία θα σας ενημερώσει γραπτός για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα αυτά και στα πρακτικά της συνεδρίασης. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της περίοδου ψηφοφορίας από τώρα μέχρι τη μισή. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης με την αλλαγή, αυτή τη μικρή αλλαγή στη σειρά των σημείων της ημερήσης διάταξης. Το επόμενο σημείο λοιπόν είναι η θέσπιση του νομικού πλαισίου για την επίτευξη της κλιματικής ιδιαιτερότητας και η τροποποίηση του κανονισμού 2018-1999, το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα. Ο νόμος για το κλίμα είναι πολύ σημαντικό θέμα. Είναι ο κρογωνίος λίθος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας η Επιτροπή ΙΤΡΗ είναι συνδεδεμένη επιτροπή στην νομοθετική διαδικασία δυνάμει του άρθρου 57 στην πολύ σημαντική αυτή πρόταση. Εν τόσο λίγο θα καλέσουμε τον εισηγητή μας τον κύριο Κρασνοντέμσκι για να μας παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης και τις 51 τροπολογίες. Έχουμε προβλέψει 35 λεπτά για την συζήτηση του σημείου αυτού Οπότε σας θερμοπαρακαλώ να είστε λακωνικοί και συγκεκριμένοι για να σεβαστούμε το χρόνο. Θα μιλήσει πρώτα ο εισηγητή για 4 λεπτά, κατόπιν οι εισηγητέ για 2 λεπτά ο καθένα. Και αν απομείνει χρόνο, θα δώσω το λόγο και στα άλλα μέλη, στου άλλου ευρωβουλευτέ που θα το ζητήσουν. Στο chat της πλατφόρμας μπορείτε να στήσετε το λόγο και θα συντάξει κατάλογο αγορητών η Γραμματεία. Αν μας μείνει και άλλος χρόνος, θα δώσω το λόγο στον τμηματάρχη από την DG Κλίμα για μια σύντομη παρέμβαση, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στο τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή για να δευτερολογήσει. Ο λόγος λοιπόν στον κύριο Κρασνοντέμσκι και τον παρακαλώ να μας παρουσιάσει σε τέσσερα λεπτά τη γνωμοδότησή του. Με βλέπετε, με ακούτε, ελπίζω. Ευχαριστώ, Κριστιαν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω κάποια ε, βασικά σημεία της γνωμοδότησής μου, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Καταρχάς, όπως όλοι συμφωνήσαμε, ε, θα πρέπει να μειωθούν δραστικά οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα και των καυσαίριων γενικώ και να έχουμε ισχυρή δράση Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Παρόλο που το πολιτικό κλίμα έχει αλλάξει τώρα και λόγω κρίση, το θέμα αυτό τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου είναι πολύ σημαντικό. Επίση, οι δράσει θα πρέπει να είναι στοχοθετημένε, αποτελεσματικέ και δίκαιε και φυσικά συμβατές με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό να επιμείνουμε σε ε, τον επικείμενο έλεγχο επιπτώσεων του κινδύνου από την μείωση αυτή που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις εθνικές ιδιαιτερότητες γιατί οι χώρες μας μέχρι τώρα έχουν στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα εθνικά σχέδιά τους αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις οικονομικές συνέπειες και τα επακόλουθα της κρίσης της πανδημίας COVID-19. Η μελέτη αυτή αντικτύπου, η μελέτη επιπτώσεων, θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα επακόλουθα της κρίσης αλλά και των μελλοντικών κρίσεων. Γιατί έχουμε τώρα την πανδημία COVID-19, αλλά ταυτόχρονα η μελέτη επιπτώσεων θα πρέπει να εκτιμήσει και την πιθανή χρηματοοικονομική υποστήριξη που θα χρειαστεί για να υλοποιηθεί ο στόχος της ουδετερότητας ε, λόγω κρίσεων. Χθε στην Ολομέλεια είχαμε το πακέτο στήριξης, ε, το σχέδιο ανάκαμψης ε, και δεν αποκλείται στο μέλλον να έχουμε και άλλες κρίσεις που θα χρειαστούν κάποιες τροποποιήσεις. Το δεν θα πρέπει δεν θα πρέπει να προεξοφλούμε την έκβαση της αξιολόγηση των επιπτώσεων, ούτε και την πιθανή αύξηση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία της γνωμοδότησής μου. Επίσης, το επόμενο σημείο αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μέχρι στιγμής, όπως ξέρουμε, όλοι οι στόχοι ε, για την μείωση των καυσέριων, συμφωνούνται σε επίπεδο Συμβουλίου με βάση και τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπισμένος ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των στόχων για το κλίμα θα πρέπει να έχουν προηγουμένως μία αξιολόγηση από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο. Συγγνώμη, αλλά έχει διακοπεί η σύνδεση με τον κύριο Κρασνοδέμσκι. Hello. Yes, we can hear you now. Κύριε Κρασονοντέμσκι, προς χάσαμε τη σύνδεση, αλλά τώρα σας ακούμε και πάλι. Οπότε δεν θα πρέπει μόνο να καθορίζουμε τους στόχους, αλλά να σχεδιάσουμε και κάποιες διαδρομές, κάποιες πορείες για την υλοποίηση. Ανάψτε και την κάμερά σας κύριε Κρασονοδέμψη, γιατί δεν σας βλέπουμε. Do you hear me? Do you see Μ' ακούτε τώρα, με βλέπετε? Σας ακούμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Εσείς μας ακούτε? I can hear you, but... You can go on without camera. Thank you. Please. Okay. Συνεχίστε χωρίς uh, κάμερα. Λυπάμαι, δεν ξέρω γιατί συνέβη αυτό. η πολιτική για το κλίμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε στόχους, αλλά και σε καθορισμό της πορείας για την υλοποίησή τους. Λυπάμαι, αλλά οι, οι παρεμβάσεις χωρίς εικόνα δεν μεταφράζονται. Should also should take into account national circumstances as energy mix, security of energy supply, employment structure, e-, economic capacities. Um,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 με την ταξινόμηση σε ETS ή εκτός ETS θα πρέπει και διάφοροι οικονομικοί φορείς να συμβάλλουν. Επίσης έχουμε εθνικές πορείες για τη μείωση των εκπομπών σε διάφορους τομείς. Ε, έτσι θα μπορέσουν και διάφοροι τομείς να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα με τον προγραμματισμό των απαραίτητων επενδύσεων. Βέβαια αυτές οι διαδρομές, αυτές οι πορείες θα πρέπει να είναι δεικτικές κατευθυντήρες γραμμές και θα πρέπει να, αναπτυχθούν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησής τους σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως είναι κάποιες κρίσεις σαν αυτή που περάσαμε και περνούμε. Το επόμενο σημείο. Προτείνω η έννοια της διαδρομής ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο προτείνω να αναβληθεί με, την, με τη μορφή κατεξοδότηση πράξεων. Η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαρακτήρισε αυτή την πρόταση ως απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβει κάποιες νομοθετικές αρμοδιότητες για να καθορίζει στόχους εκπομπών. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι η νομική μας υπηρεσία διαπίστωσε ότι η θέσπιση αυτής της διαδρομής, της πορείας προς το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, στην ουσία σημαίνει καθορισμό της διαδρομής προς μια κλιματικά ουδέτερη κοινωνία και οικονομία. Ενώ η διαδρομή, το trajectory αυτό, είναι ουσιαστικό στοιχείο ε, της υιοθέτηση που δεν χωρείται όμως ε, ε, η χάραξή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να το λάβει αυτό υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να μην το δεχτεί. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, και λυπάμαι που δεν μπόρεσα να συνδεθώ και με εικόνα, ε, θέλουμε μελέτη επιπτώσεων, ρόλο του Συμβουλίου ε, στις ε, διαδρομές αυτές, ε, όλων των τομέων της οικονομίας και το θέμα των κατεξουδότηση πράξεων, που θα πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία της γνωμοδότησής μου και σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κραστοντεύσκη. Περάμε αμέσω στους σκιώδεις γιατί έχουμε πολύ σημαντικά θέματα και λίγο χρόνο σήμερα. Ο κύριος Πίπερ που είναι παρόν στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ε, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε θα μιλήσω στη μητρική μου γερμανικά. Θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή, τον κύριο Κρασνοντεύσκη, για την πρόταση αυτή που τη βρίσκουμε πολύ καλή και ε, ευπρόσδεκτη. Έχει καλές προτάσεις, ας πούμε μια προσέγγιση ουδέτερη προς την τεχνολογία, αναφέρεται βεβαίως και στην κρίση του COVID-19 και χρειάζεται εκεί προσαρμογές. Νομίζουμε ότι με τις καταξιοδότηση πράξης δεν γίνεται δουλειά, χρειάζεται κανονική νομοθεσία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επίσης θεωρούμε ότι αν θα χρειαστεί να επαναξιολογηθεί ε, ο στόχος του 2030, αυτό θα πρέπει να γίνει με μελέτη αντικτύπου και όχι ε, να έχουμε μία πτήση στα τυφλά, χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνουμε και χωρίς πηξίδα. Δεν προτείνουμε εμεί τώρα νέα ημερομηνία για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση, αλλά θα μπορούσα να φανταστώ το ΕΛΚ να ζητήσει ρητά και κατηγορηματικά να γίνει μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων. Και ενδεχομένω να αφήσουμε ανοιχτό το θέμα το χρονικό. Ακόμα είναι υποσυζήτηση αυτό στην ομάδα μας. Θα σταματήσω εδώ. Μια καταληκτική παρατήρηση μόνο. Θα επιθυμούσα πάρα πολύ, κύριε Σιγητά, να ήσασταν λίγο πιο αισιόδοξο, να έχετε έτσι λίγο μεγαλύτερη εφορία και πιο θετική διάθεση για την προστασία του κλίματος, γιατί και αυτές οι επενδύσεις είναι τεράστια ευκαιρία για τη βιομηχανία, Υπάρχει ε, πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτή την τεχνολογία και μπορούμε πολύ καλύτερα να λειτουργήσουμε έτσι. Και αυτό θα ευνοήσει και την οικονομική ανάπτυξη Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Βιομηχανίας, είμαι και λίγο στεναχωρημένος και λυπημένος. Εδώ κατά 80% είναι, είναι θέματα ενεργείας. Και εμεί είμαστε η Επιτροπή Αρμόδια για την Ενέργεια και καθήλυνα αρμόδια επί δηλαδή είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος στο Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα ενέργειας, είναι δική μας αρμοδιότητα και όχι της ΕΜΒΗ. Ευχαριστώ πολύ, σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Γκονζάλης Κασάρες. Γεια σας, μ' ακούτε, εντάξει. Θα συνεχίσω στα ισπανικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ορόσημο για την ε, κλιματική ουδετερότητα στην Ευρώπη το 2030. Επίσης, εχθές ζήσαμε μια ιστορική στιγμή με την πρόταση του σχεδίου ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναθέρμανση τη οικονομία και με αυτή την νομοθεσία και την πρόταση για άλλη μια φορά η Ευρώπη δείχνει πόσο είναι προσιλωμένη στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή και υπέρ τη πράσινη ανάκαμψη και του πράσινου συμφώνου. Ωστόσο, η πρόταση χρειάζεται προσαρμογή τουλάχιστον σε αυτά που ζητάει το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν περισσότερα μέτρα και περισσότερα μέσα που προσφέρονται για να είμαστε αποτελεσματικοί στη δράση μας. Αυτό είναι δική μας δουλειά να γίνει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κρασνοντεύσκη για το σχέδιο πρότασής του. Έχει θετικά στοιχεία και εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν να φτάσουμε στο στόχο μας της κλιματικής ουδετερότητας με δίκαιο τρόπο και χωρίς να μείνει κανένας ε, στο περιθώριο. Παρ' όλα αυτά, γιατί έχει βγει ένας στόχος για το 2030. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν ξεκινούν όλα τα κράτη-μέλη από την ίδια αφετηρία, ότι έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Θα πρέπει να έχουμε και το μηχανισμό δίκαιης μετάβασης. Είναι σημαντικό ο στόχος της κλιματικής ουτερότητας να είναι και εθνικός. Αν δεν είναι κάτι τέτοιο θα υπάρξει κίνδυνος να ανοίξει η ψαλίδα για διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και θέλω να ρωτήσω, τι τεχνολογίες θέλετε να υποστηρίξετε ε, ως προς την κλιματική ουδετερότητα και είναι αυτές συμβατές με την ταξινόμηση των στόχων και των προτεραιοτήτων. Από το Ρινιού, ο κύριος Φέντερλε. Σας ευχαριστώ κύριε Καζανοντεύσκη για το σχέδιο έκθεσης. Έχουμε κάποια κοινά σημεία όταν μιλάμε για μια προσέγγιση ουδέτερη ως προς την τεχνολογία και κλιματικά ουδέτερη. Όμως το επίπεδο φιλοδοξίας διαφέρει λίγο σε σχέση με αυτό το οποίο θα ήθελε να δει το Renew Europe. Υπάρχει τώρα η ευκαιρία δεδομένης της κρίσης να φροντίσουμε να επανεκκινήσουμε την οικονομία και την κοινωνία με έναν τρόπο πιο προοδευτικό στα κλιματικά. Έχουμε τους στόχους για τις εκπομπές, κλιματική ουδετερότητα για κάθε κράτος μέλος, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω από αυτήν την πράσινη μετάβαση. Όπως ε, και το ΕΛΚ θέλουμε και εμείς μια πιο θετική προσέγγιση για το μέλλον, γιατί γνωρίζουμε ότι έχουμε μια νέα ευκαιρία για την οικονομία της Ευρώπης. Η ρύθμιση λοιπόν αποτελεί τον βασικό πυλώνα για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας, αλλά θα πρέπει η Επιτροπή μας να τονίσει την ανάγκη της έρευνας τεχνολογίας, των δυνατότητων απορρόφησης άνθρακα για να επιτύχουμε την κλιματική ουδετερότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Σας ευχαριστώ κύριε Φέντερλε. Ο κύριος Μπουκχάιτ δεν έχει συνδεθεί, αντιλαμβάνομαι, ο σκιώδης ηγητής της ομάδας ID. Αν συνδεθεί, ειδοποιήστε μας. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπλος από τους Πράσινους. Κύριε Μπλος. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κρασνοντεύσκη για το σχέδιο αυτό. Χτες νομίζω είχαμε μια ιστορική στιγμή στην Ευρώπη. Θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση του ιού και πραγματι υπάρχει ένα θετικό πνεύμα το οποίο πρέπει να προληφθεί και από την κλιματική νομοθεσία για να μπορέσουμε να πούμε ότι θα σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή και να διατηρήσουμε τις δουλειές και να διατηρήσουμε την βιομηχανία στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κάνει η σχετική νομοθεσία. Και φέτος είχαμε κλιματική κρίση, είδαμε διάφορες ξηρασίες ακόμα και στην Πολωνία Οπότε πρέπει να ακούσουμε τα όσα μας λέει η επιστήμη και να μπουν επιστημονικοί στόχοι. Το σκεπτικό της Κομισιόν είναι να υπάρξει μια νομοθεσία ε, που θα δίνει κάποιες κατευθύνσεις για το κλίμα και μετά να δούμε τα ενεργειακά συστήματα και τους διάφορους κλάδους. Νομίζω αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε εδώ. Και επίσης βεβαίως η Ήτρε σχετίζεται και με το άρθρο 57, το άρθρο 10. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να επηρεάσουμε την διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο νόμος αυτός να αποτελέσει την βάση για την ενημέρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Οπότε η αναβολή της διαδικασίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Επίσης, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να υποτασσόμεθα στο Συμβούλιο. Είμαστε αιρετοί και πρέπει να προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις αυτόνομα. Λοιπόν, ας είμαστε λοιπόν επιτυχείς για τη βιομηχανία, για το κλίμα, για την ενέργεια. Κάθε κρίση πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κρίση. Και με τον νόμο αυτό νομίζω μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μπλος. Τελευταίος. Από, τελευταία από τους σκιοδησηγητές, η κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον εισηγητή. Νομίζω έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με διαφορετικές απόψεις βεβαίως. Νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το θέμα. Πάρα πολλά εξαρτώνται από αυτή την νομοθεσία, πρέπει να το πούμε. Πρέπει να συνδεθεί η ανοικοδόμηση στην Ευρώπη με τους κλιματικούς στόχους. Αλλιώς ε, θα χάσουμε την ευκαιρία και δεν μπορούμε να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το πούμε. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια θαραλέα απόφαση για να γίνει η αρχή. Να έχουμε δηλαδή τους στόχους μέχρι, τους, ε, μέχρι το 2030 δεν μας ικανοποιούν αυτοί, πρέπει να είναι ακόμη υψηλότεροι, όπως ε, άλλωστε θα προτείνουμε και με τις τροπολογίες μας. Επίσης ε, υπάρχουν διάφοροι κλάδοι που μπορούν να εισαχθούν, κατά οποίο μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς ε, να μην συνεισφέρει. Επίσης για την τεχνολογική ουδετερότητα πρέπει να συζητήσουμε. Επί της αρχής λέμε θα πρέπει βεβαίως ε, όσοι ε, ρηπαίνουν να υπομισθούν το κόστος ανακύκλωσης και των σχετικών και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να ανοίξει η πόρτα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εις βάρος των ορυκτών καυσίμων τα οποία επιδοτούνται εδώ και χρόνια. Και πρέπει να συζητήσουμε βεβαίω και το θέμα των πράξεων καταξιοδότηση και των εθνικών μέτρων. Εδώ πέρα συμφωνούμε με τον εισηγητή, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι εννοεί εδώ πέρα. Άρθρο 10, ναι, θετικό. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να έχουμε ο στόχο την κλιματική ουδετερότητα που θα συνδεθεί με την Συμφωνία των Παρισίων, αλλιώς δεν θα προχωρήσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια θαραλέα ε, νομοθεσία. Σας ευχαριστώ κυρία Ένστ. Δεν ε, έχουμε λάβει κάποιο συγκεκριμένο αίτημα για το KHDI. Και ο εκπρόσωπος Κομισιόν δεν έχει συνδεθεί. Τέλο πάντων, θα έχουμε και άλλη ευκαιρία. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Είναι στην αίθουσα ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν. Α, μάλιστα. Ε, μου είπαν ότι δεν ήταν παρόν. Α, είναι στην αίθουσα λοιπόν, γι' αυτό δεν φαίνεται συνδεδεμένος. Οπότε θα δώσω λόγο στον κύριο Λούκα Ντεκάρλη, προϊστάμενο στην DG Σας ευχαριστούμε κύριε Μπουσόη και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστούμε και τον εισηγητή, το συντάκτη γνωμοδότη και του σκιώδη εισηγητέ για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το νόμο για το κλίμα, που είναι σημαντικό νομοθέτημα. Τώρα, βέβαια, έχουμε εστιαστεί στην κρίση του COVID, αλλά δεν θα πρέπει να μελήσουμε την ανάγκη μετριασμού των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει λοιπόν και να προστατεύσουμε την κοινωνία, αλλά και να ενισχύσουμε τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν θα, χρω... δεν θα μακρηγορήσω, θα ήθελα απλώς να μιλήσω για τη δημοκρατική διαδικασία και τη θέσπιση των στόχων. Στο νόμο για το κλίμα ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ε, τους δύο συνομοθέτες, να θέσουν στην νομοθεσία τους στόχους ε, για την υλοποίηση της, τεχνική, της κλιματικής ουδετερότητας συνολικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το 2050. Και οι συνομοθέτε υλοποίησαν ε, και τους στόχους, ε, μάλλον όχι, έθεσαν του στόχου και το 2030 και θα πραγματοποιήσουμε αξιολόγηση. Τώρα δεν ξέρω πόσο στις μελέτες επιπτώσεων θα λάβουμε υπόψη και τα επακόλουθα του COVID-19. Πριν από δύο εβδομάδες ε, είχαμε ε, υποβάλει μια πρόταση και φυσικά δεν έχουμε ακόμη πλήρη δεδομένα για την παρούσα οικονομική κατάσταση λόγω της κρίσης. Άλλωστε, ε, θα έχουμε και μελέτη για το 2030, όχι για δύο-τρει μήνε από τώρα. Σε ό,τι αφορά τι πορείε ή τι διαδρομέ, δεν ήταν στόχο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σφετεριστεί οποιαδήποτε εξουσία από του συνομοθέτε. Οι συνομοθέτε, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο έχουν την ε, εξουσία να υποβάλουν τους στόχους και τις ε, διαδρομές. Το θέμα των διαδρομών δεν ήταν να θέσει στόχους, αλλά να δώσει ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της πρόοδου στην προσπάθεια επίτευξη κλιματικής ουδετερότητα. Υπό αυτό το πνεύμα πιστεύαμε και κρίνουμε ακόμη ότι είναι κατάλληλο εργαλείο η καταξιδότηση πράξη. Ο στόχος, ε, ο στόχος είναι το σημαντικό, όχι τα μέσα. Και ήταν σημαντικό αυτό ε, να το συζητήσουμε με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το καλύτερο μέσο για την υλοποίηση των στόχων που έχουν θεσπίσει οι συνομοθέτες. Ευχαριστούμε κύριε Λούκα Ντεκάρλη. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και επανέρχομαι στον εισηγητή μας, τον κύριο Κρασναντέμσκι, που σε ένα-ενάμιση λεπτό θα πρέπει να απαντήσει ε, στα σχόλια ή στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Παρακαλώ κύριε Κρασνοντέμσκι. Ελπίζω να με βλέπετε τώρα και να με ακούτε. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι δεν έχουμε μεγάλες διαφορές μεταξύ μας. Έχουμε αρκετή συμφωνία, γιατί όλοι θέλουμε να υλοποιήσουμε τους κλιματικούς μας στόχους και την κλιματική ουδετερότητα. Το θέμα είναι πώς, με ποιο τρόπο, με ποια εργαλεία, με ποια μέσα. Αυτό που θα ήθελα να πω στη γνωμοδότησή μου πρώτα απ' όλα είναι ότι θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Γιατί όπως γνωρίζουμε τώρα, αλλά και που, κάτι που ισχύει γενικά, μπορεί να συμβεί ανα πάσα στιγμή κάτι απροσδόκητο. Και θα κληθούμε να το λάβουμε υπόψη, οπότε θέλουμε και μελέτη αντικτύπου. Συγκεκριμένη, αλλά και αρκετά ευρεία, περιεκτική. Και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σχόλιο κάποιων συναδέλφων, ότι η Ευρώπη έχει δύο και τα σημεία φετηρίας των χώρων μελών πολλές φορές είναι διαφορετικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη συζήτηση κάποιους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Για να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά σημεία κίνησης και τις διαφορές των εθνικών ενεργειακών σχεδίων. Επίσης, δεν θα πρέπει να, προεξοφλούμε την έκβαση, τα αποτελέσματα της μελέτης επιπτώσεων. Και δεν θα πρέπει ήδη από τώρα να θεσπίζουμε αύξηση των στόχων μείωσης των εκπομπών, αύξηση των ποσοστών της μείωσης. Είναι πολύ νωρίς να το προδικάζουμε από τώρα. Καλό είναι να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά όχι υπερβολικά φιλόδοξοι. Γιατί είναι μεγάλο το εύρος της φιλοδοξίας, η ψέλιδα της φιλοδοξίας. Μερικές φορές η υπερβολική φιλοδοξία είναι αντιπαραγωγική. Το ζητούμενο είναι να υλοποιήσουμε τους στόχους. Και θα το κάνουμε όντας ρεαλιστική και ελαστική και ευέλικτη. Επίσης, λέω στην γνωμοδότησή μου ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τους επιμέρους τομείς. Γι' αυτό θέλω περιεκτική και γενική ευρεία αξιολόγηση επιπτώσεων. Αν δούμε τη συμβολή κάθε τομέα στην μείωση των εκπομπών, βλέπουμε τα διαφορετικά επίπεδα. Σίγουρα ο ενεργειακό τομέα παράγει τι περισσότερε εκπομπέ. Αλλά ο ενεργειακό τομέα είναι αυτό που έκανε και τι πιο φιλόδοξε προσπάθειε και τις πιο μεγάλες προσπάθειες για τη μείωση. Ας μην λοιπόν ε, παραμελούμε τους υπόλοιπους τομείς και τη συμβολή τους. Και θα πρέπει οι κατευθυντήριες γραμμές να τίθενται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ως προσανατολισμός όμως, ως κατευθυντήριες γραμμές και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με τη βιομηχανία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τώρα έρχομαι στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λέω ότι θα πρέπει όλοι οι στρατηγικοί στόχοι να συζητούνται μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Η θέσπιση τους θα, θα πρέπει να γίνεται και από, τους, από τα δύο θεσμικά όργανα. Και χθε είδαμε στην πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης ότι η στρατηγική απόφαση δεν ελήφθη από το Συμβούλιο. Άρα το ψήφισμά μας δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου. Και γι' αυτό είμαι κατά των κατεξοδότηση πράξεων τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί θέλω να εμπλέξω περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας, θα πρέπει να συνεργαστούν και τα τρία θεσμικά όργανα μεταξύ τους. Χωρίς να μελούμε το σημαντικό ρόλο που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει τη διαδικασία. Επίση, δεν μπορούμε να αλλάζουμε μια στρατηγική χωρίς τη συνένεση, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με το Συμβούλιο. Και αυτό το τονίζω στην γνωμοδότηση. Γενικώ, λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να κοιτάξουν και να μελετήσουν πιο διεξοδικά την γνωμοδότησή μου. Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξο ότι θα βρούμε συμβαστικές λύσεις, γιατί ως Επιτροπή είμαστε αρμόδιοι και για τη βιομηχανική πολιτική και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη βιομηχανική πολιτική στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Κρασνοντέμσκι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κρασνοντέμσκι και για την παρουσίασή σας και για την έκθεσή σας. Είναι πολύ σημαντικός ο στρατηγικός στόχος του 2050 και ανάγκη να ορίσουμε ένα ενδιάμεσο στόχο για το 2030. Περιμένουμε μια γερή μελέτη αντικτύπου ε, στην οικονομία, στην απασχόληση, ε, στην ανταγωνιστικότητα, στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ε, και πώς μπορούν τα διάφορα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν, σεβόμενοι πάντα τις εξουσίες και τα προνόμια του κάθε θεσμικού όργανου. Προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. 5η 4 Ιουνίου στι 12 το μεσημέρι, δηλαδή σε μια εβδομάδα από τώρα. Θα ήθελα απλώ να σα θυμίσω, συνάδελφοι, ισχυρέ συστάσει που μέχρι τώρα τι ακολουθούσατε όλοι σα να καταθέσετε τις τροπολογίες σας όσο γίνεται στα αγγλικά. Και επίσης, αν γίνεται, εξ ονόματος πολιτικής ομάδας ή κάποιος να συνυπογράφει από την πολιτική σας ομάδα, η μερικα μέλη, τουλάχιστον τέσσερα, της ομάδας σας. Αυτό θα μας βοηθούσε. Μέχρι τώρα ε, έχουμε λειτουργήσει πολύ καλά με αυτές τις τάσεις. Ευχαριστώ πολύ και θα επανέλθουμε, είμαι βέβαιος, ε, όταν θα έχουμε τις τροπολογίες και πριν την ψηφοφορία που προβλέπεται για το Σεπτέμβριο. Στη Δε Ολομέλεια θα πάει ε, τον Οκτώβριο, στην πρώτη Ολομέλεια το Οκτώβριο. Εξαρτώμεθα από το χρονοδιάγραμμα και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είμαστε κάπου στη μέση, ε, ένα συμβιβασμό έχουμε βρει ανάμεσα στη δική τους αρχική και τη δική μας αρχική θέση. Είναι πολύ σημαντική πάντως αυτή η νομοθεσία και θα πρέπει να προχωρήσει. Πάμε στο επόμενο θέμα, όπως αλλάξαμε την μέρη διάταξη, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, μια νέα στρατηγική, βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Η συγκητής είναι ο κύριος Καλέντα, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι το Νοέμβριο του 2019 αποφάσισε ήδη η Επιτροπή μας να ε, καταρτήσει μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας για ε, το μακροπρόθεσμο βιομηχανικό μέλλον της Ευρώπης. Στη συνέχεια στις 10 Μαρτίου, θυμάστε ότι συζητήσαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ε, ανακοίνωσή της, η οποία ήταν μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη. Με τις συνέπειες του COVID-19 και τη σχετική κρίσης στην ευρωπαϊκή βιομηχανία, θέλουμε να αναπροσαρμόσουμε τη θέση μας ε, και να λάβουμε υπόψη αυτές τις συνέπειες. Ε, εξού και η στρατηγική αυτή, η οποία θα λάβει υπόψη τις νέες πραγματικότητες, ε, την επίπτωση του COVID, τις οικονομικές συνέπειες αλλά και το σχέδιο ανάκαμψης που πρότεινε χτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η νομοθεσία λοιπόν και να λάβουμε θέση για τη στρατηγική της Ευρώπης, να χαράξουμε και εμείς στρατηγική γι' αυτό. Θα κάνουμε μια πρώτη συζήτηση τώρα, 35 λεπτά μόνο, ε, φυσικά θα επανέλθουμε και σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να θυμίσω ότι έχουμε ήδη συζητήσει μερικά από τα στοιχεία αυτά με τον Επίτροπο Μπρετών και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ντομπρόφσκης σχετικά πρόσφατα. Είμαστε σε συνεχή διάλογο και θα ε, συνεχίσουμε να το συζητάμε με σημαντικούς επιτρόπους. Ε, ισχύουν οι ίδιοι οι κανόνες. Πρώτα θα ακούσουμε τον εισηγητή, μετά το σκιώδη. τέσσερα λεπτά ο κύριο Καλέντα, δύο λεπτά οι σκιώδη εισηγητές και μετά ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και αν έχουμε χρόνο. Ζητήστε το λόγο για σύντομε παρεμβάσει στο ΚΑΤΣΙΑΙ. Το λόγο έχει αμέσω ο κύριο Καλέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ε, πρόκειται πραγματικά για μια ομαδική προσπάθεια με τους ε, αγαπητούς ε, συνεισηγητές και είχαμε και την ευκαιρία να συναντηθούμε και με την Αρμόδια Επίτροπο σε μια πάρα πολύ παραγωγική συνεδρίαση για να αντιληφθούμε την κατάσταση των οικοσυστημάτων. Τώρα, αν μου επιτρέπετε, θα μιλήσω Ιταλικά. Το έγγραφο το οποίο έχετε λάβει είναι οργανωμένο σε δύο φάσεις γιατί η κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά με τον κορονοϊό. Οπότε, ενώ οι στόχοι της ε, ψηφιοποίησης και του περιβάλλοντος ε, παραμένουν απολύτως οι ίδιοι, πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, μια οικονομική κρίση η οποία θα προκαλέσει μια ύφεση του 7,4% σύμφωνα με τις προβλέψεις ε, που ε, δεν έχει προηγούμενο στο πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, αυτό θα κρίνει δύο φαινόμενα. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε μία μείωση των διαθέσιμων κεφαλαίων για επενδύσεις των επιχειρήσεων και το δεύτερο φαινόμενο θα είναι μία ανισορροπία στο εσωτερικό της ε, εσωτερικής αγοράς ε, όσον αφορά την στήριξη ε, που δίνεται από τα κράτη-μέλη όσον αφορά το πλαίσιο των προσωρινών κρατικών ενισχύσεων. Οπότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα ε, στην πρώτη φάση της ανάκαμψης με το θέμα της ισορροπίας της εσωτερικής αγοράς και είναι σημαντικό για εμάς στο μέτρο του δυνατού τα ταμεία του New Generation Fund ε, να χρησιμοποιηθούν και για προγράμματα ευρωπαϊκά που θα διαχειρίζεται η Κομισιόν. Νομίζω αυτή η ανισορροπία ε, θα, θα αποκατασταθεί σε έναν βαθμό. Δεύτερον, έχουμε το θέμα της ε, σχέσης μεταξύ ε, χρέους και μετοχικού κεφαλαίου. Χάρη στα προγράμματα ρευστότητας θα έχουμε πολύ περισσότερο χρέος στις επιχειρήσεις και λιγότερα άρα κεφάλαια προς επένδυση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε το τι θα γίνει με το μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Να θυμάστε επίσης πως έχουμε δύο μεταβάσεις, ψηφιακή και περιβαλλοντική, που απαιτούν πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Επίσης, αυτό το οποίο είναι ταυτόχρονα σημαντικό είναι να έχουμε μια τότε να αμυνθούμε σε λαθασμένες συμπεριφορές στο διεθνές επίπεδο, να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις εξαγορές και της μετατόπισης της ε, παραγωγικής αλυσίδας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων δεν θα διαβάσω ολόκληρο το έγγραφο το οποίο έχετε λάβει. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι η δεύτερη φάση αφορά τον μετασχηματισμό και η διαχείριση ε, αυτό του μετασχηματισμού σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μέσα τα οποία θα λειτουργούν και σε αυτό θα επικεντρωθούμε και όχι στη θεωρία. Οπότε, παραδείγματο χάρη, να χρησιμοποιηθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να μπορέσουμε να φτιάξουμε σχήματα οικονομικά, αλλά και να έχουμε ένα σύστημα δίκτων απόδοσης και performance indicators, το οποίο θα είναι σοβαρό. Και τέλος, έρχομαι στο τελευταίο. Πρέπει να προχωρήσει το θέμα το περιβαλλοντικό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε σίγουροι με βάση μια ανάλυση αντικτύπου ότι ειδικά στη φάση της ανάκαμψης δεν θα υπομιστούν οι επιχειρήσεις άλλα βάρη πέρα από αυτά τα οποία ήδη ε, έχουν λόγω της κρίσης του COVID. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλέντα. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Και πράγματι έχετε δίκιο, είναι ομαδική εργασία γιατί έχουμε μια στρατηγική θέση της ε, Επιτροπής μας. Όπως είπαμε πάμε τώρα γρήγορα στους κοιόδης εισηγητές. Δύο λεπτά για τον καθένα έχουμε ενδεικτικά. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ τον κύριο Μπέρντσεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή ο οποίος ε, πράγματι ε, έχει συνεργαστεί πάρα πολύ καλά μαζί μας. Έχουμε πολλά θετικά πράγματα στην έκθεση. Έχουμε κάποια πράγματα τα οποία θα θέλαμε να συζητήσουμε και θα προτείνουμε ως ΕΛΚ και κάποιες δικές μας ιδέες. Τώρα, σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι απαιτείται ένα πάρα πολύ ισχυρό μήνυμα στην βιομηχανική στρατηγική από την Επιτροπή μας, γιατί η βιομηχανία είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και θα είναι και η ραχοκοκαλιά της ανάκαμψης. Ε, κοιτώντας λοιπόν το πακέτο ανάκαμψης που προτάθηκε χτες, θεωρούμε ότι απαιτείται και ένα ισχυρό μήνυμα από την Επιτροπή μας ακριβώς για να διαμορφώσει την ιδέα της στρατηγικής αυτονομίας. Επίσης, ε, η κρίση κατέδειξε ότι εξαρτώμεθα υπερβολικά από άλλα μέρη του κόσμου, οπότε πρέπει να επανέλθει η παραγωγή στην Ευρώπη, όπου αυτό είναι δυνατό, να προστατεύσουμε τις εταιρείε απέναντι σε κρατικά στηριζόμενες εταιρείες τρίτων χωρών, απέναντι σε εχθρικές εξαγορές, να επενδύσουμε στην αλυσίδα υπεραξίας, αυτό το οποίο η κομισιόν και να επενδύσουμε στις υποδομές που θα βοηθήσουν τη βιομηχανία μας να κάνει την ενεργειακή μετάβαση. Πρέπει όμως κυρίως να δούμε την καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη γιατί πρέπει να φροντίσουμε και άλλε μέρη του κόσμου να εξαρτώνται από εμάς. Άρα να είμαστε καινοτόμοι και για να έρθουμε στο πακέτο της ανάκαμψης. Αν αρχίσουμε να δανειζόμαστε λεφτά από τις επόμενες γενιές, πρέπει να τα επενδύσουμε στην ενίσχυση της οικονομίας. Και βεβαίω η βιομηχανία μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία ως προς αυτό. Θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και ως ΕΛΚ θέλουμε να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους άλλους κοιόδης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέρενσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπέρασεν. Ερχόμαστε στο σκιώδη από την ομάδα Ρινιού, ο κύριος Μπρούντνερ. Ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Καλέντα για το εξαιρετικό σχέδιο εκθεσής του και για την εξαιρετική συνεργασία του με τους συναδέλφους και οδησηγητές. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η έκθεση για το μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει στεναρή όσο και καθαρή θέση γι' αυτό θα πρέπει επιγόντως να σώσουμε ε, τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία μας από την πρωτοφανή κρίση, να έχουμε ανάκαμψη πράσινη, καινοτόμα, χωρίς αποκλεισμούς και κυρίαρχη. Βεβαίως χαίρομαι ε, ε, με το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκε χθες. 500 δισεκατομμύρια επιχορηγήσεις, 433 τύπου ΕΣΠΑ ε, και τα 67 υπόλοιπα δισεκατομμύρια επιχορηγήσεων θα γίνουν με κλασικό πρόγραμμα. Αυτό είναι μια απτή ε, απόδειξη αλληλεγγύης. Αλλά δεν θα πρέπει μόνο να ε, σώσουμε τη βιομηχανία από τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε μεγάλα κοινά ευρωπαϊκά σχέδια και να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες. Για παράδειγμα, να ενισχύσουμε το διαστημικό πρόγραμμα για να έχουμε ένα αστερισμό ευρωπαϊκών δορυφόρων και να εξασφαλίσουμε την ψηφιακή μας κυριαρχία. Ε, η ανάκαμψη της οικονομίας δεν ε, χρειάζεται μόνο χρηματοδότηση, χρειάζεται και ένα πλαίσιο πιο ευνοϊκό, ρυθμιστικό. Ε, για Να ενισχύσουμε τα μέσα οικονομικής προστασίας και άμυνας, κανόνες ανταγωνισμού και να υιοθετήσουμε μια ευρωπαϊκή προτιμησιακή ρήτρα στις ε, δημόσιες προμήθειες στρατηγικού χαρακτήρα ε, για την παραγωγή επίση και ε, των πρώτων υλών. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επαναπατριστούν οι στρατηγικές βιομηχανίες στην Ευρώπη. Τίποτα δεν πρόκειται να είναι όπως ήταν στο παρελθόν. Ελπίζω αυτή η κρίση να αφύπνισε την αλληλεγγύη αλλά και τις δυνάμεις μας για συνεργασία και αγωνιστικότητα για να είμαστε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην υπηρεσία των πολιτών. Ευχαριστώ τους συναδέλφους των πολιτικών ομάδων και τον εισηγητή φυσικά για να προχωρήσουμε προς μια πραγματική ανάκαμψη της βιομηχανίας στην Ευρώπη, φιλόδοξη, αλληλέγγυα και ενάρετη. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πάλο Μπορζία που είναι στην αίθουσα νομίζω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κάρον. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για αυτό το σχέδιο έκθεσης. Είναι πολύ καλύτερο από ότι το τελευταίο σχέδιο που είχαμε δει. Ε, θα ήθελα να χωρίσουμε την έκθεση σε δύο τμήματα. Πραγματικά αυτό το κάνει ο εισηγητής και είναι εύκολο να ε, έχουμε μια εικόνα στη στρατηγική μας μετά την κρίση. Ο εισηγητής έχει ε, πολύ θετικές προτάσεις και σημεία ε, θέλει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική παγκοσμίω, να προωθηθεί ε, ο βιομηχανικός τομέας και το φυσικό αέριο και το υδρογόνο θεωρείται ε, τεχνολογία αιχμής. Επίσης, προστατευτικά μέτρα προτείνονται, όπως είναι ο φόρο για το διοξίδιο του άνθρακα στα σύνορα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στα θεμέλια τη στρατηγική ανάκαμψη που θα ακολουθήσουμε και χαίρομαι που έχουμε συμφωνία μεταξύ όλων τους και σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά μέσα συμφωνώ με τον εισηγητή να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην είναι δάνεια αυτή η χρηματική υποστήριξη, γιατί θα έρθουμε να ε, προσθέσουμε χρέος στο χρέος, που είναι ήδη χρεωμένες επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο εισηγητής, ιδιαίτερα για τις Πράσινε. νέε θέσει εργασία. αυτές δεν θα αντικαταστήσουν ένα προ ένα όλες τις χαμένε θέσεις στη βιομηχανία. Ε, θα αλλάξει η αγορά εργασία που διέρχεται κρίση αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικά τα στοιχεία, τα τόνισα και στι δικές μου ε, τροπολογίες για την έκθεση για τη δίκαιη μετάβαση και το αντίστοιχο ταμείο. Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά. Νομίζω δεν είναι τώρα η ώρα να ζητήσουμε από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, να εφαρμόζουν επιπλέον απαιτήσει για το περιβάλλον. Εδώ αγωνίζονται να επιβιώσουν και αγωνιούν. Αυτό μπορεί να πάει σε δεύτερη φάση ε, ε, της έκθεσης για να έχουμε στην πρώτη φάση μια ευελιξία στην ανάκαμψη. Χαίρομαι για τη μελέτη αντικτύπου και επιπτώσεων που ζητάει ο ο εισηγητή για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει ε, πριν καταθέσουμε οποιαδήποτε νέα νομοθετική πρόταση. Ευχαριστώ κύριε Μπόρκια. Ο κύριος Μπλος, επίσης και όδης από πλευράς Πρασίνων για το θέμα αυτό. Γεια σας. Ελπίζω να μ' ακούτε. Ε, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ και Καλέντα για την έκθεση αυτή. Είναι πιστεύω καλή και κινείται σε καλό πνεύμα. Είναι δύσκολος ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας και χρονοβόρος, ιδιαίτερα σε τέτοιους καιρούς κρίσης που ζούμε. Και είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε από σήμερα. Είναι μια τεράστια ευκαιρία και θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Πράσινης Συμφωνίας και του Σχεδίου Ανάκαψης για να έχουμε ε, μια ουδέτερη βιομηχανία ως προς το κλίμα. Δεν είναι αυτός σκοπός ο μετασχηματισμός της βιομηχανίας. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες, ε, το περιβάλλον και να διατηρήσουμε την κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη και τις θέσεις απασχόλησης. Είναι μια τεράστια κρίση για όλη την ανθρωπότητα η κρίση του COVID. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να επικεντρωθούμε και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα Ξέρω ότι μιλάτε για το υδρογόνο και το φυσικό αέριο, ε, ε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει η κυκλική οικονομία που είναι προτεραιότητα, ε, οι φιλικές πηγές, η ηλιακή ενέργεια ας πούμε, που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας. Μπορούμε να παράγουμε ηλιακά πάνελ φωτοβολταϊκά εδώ στην Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον νεολικό κλάδο. Ε, έχει τεράστια ε, ε, δυνατότητα, είναι μεγάλο το δυναμικό. Αντλίες θερμότητας, να μην τα αναφέρω όλα, αυτά που θα μας βοηθήσουν να ανακάψουμε και να διατηρήσουμε την ευημερία μας. Θα πρέπει να ενταθεί η παραγωγή για σωστές κατασκευές, με ανανεώσιμο ε, τρόπο ηλεκτροδότησης και σε ό,τι αφορά τα εργοστάσια χάλιβα και χημικά θα πρέπει να αλλάξουν τακτική, να αλλάξουν τρόπο και τώρα να επενδύσουν στην παραγωγή με μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Πώς θα γίνουν αυτά πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρωτοπόρες αγορές ε, με προδιαγραφές για τα προϊόντα, με ειδικά εργαλεία, ε, με διαφορετικό τρόπο δημοσίων συμβάσεων και Στα, τελευταία, στα επόμενα 10 χρόνια θα πρέπει 70 εκατομμύρια νοικοκυριά και ε, κατοικίε ε, να έχουν εξοπλιστεί με φωτοβολταϊκά έτσι ώστε να είναι ουδέτερα ως προς ε, την κατανάλωση ενέργειας. Θα πρέπει να υπάρχει ένα παρατηρητήριο ε, ουδέτερο που να εποπτεύει και να παρακολουθεί τις επενδύσεις, έτσι ώστε η βιομηχανική πολιτική να μην ε, χειραγωγείται για να δημιουργούνται στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά να βρίσκουμε λύσεις τραμμένες προς το μέλλον. Αν το κάνουμε αυτό θα είμαστε σε μια μοναδική θέση. Θα είμαστε πρωτοπόροι, ουδέτεροι στο κλίμα με τεχνολογίες που αναπτύσσονται και παράγονται στην Ευρώπη. Μιλάμε για ψηφιακή επανάσταση. Α γίνει τώρα η Ευρώπη η επανάσταση ε, η βιομηχανική που θα ξεφύγει από τον άνθρακα. Ο κύριο Τομπισόφσκι, ο σκιώδη ηγητή από το ΕΣΥΑΡ. Κυρίε και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή τον Κάρλο Καλέντα για τις τους, την προσπάθειά του και την αξιόλογη έκθεσή του. Σε πολλά σημεία συμφωνώ με τον εισηγητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα προσαρμόζεται στις τρέχουσες συνθήκες και θα επικεντρωθεί σε δύο διαφορετικά στάδια. Σε στην πρώτη φάση που είναι η ανασυγκρότηση της οικονομίας και στη δεύτερη φάση που είναι η, ο μετασχηματισμός της ε, οικονομίας και της βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις ε, όχι μόνο αναγκάζονται να αναπροσανατολίσουν τις ε, επενδύσεις τους στον εξυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος, αλλά όταν δίνουν μάχη να επιβιώσουν στην αγορά με τη μείωση της παραγωγής, με την απόλυση τμήματος του προσωπικού, απόλυση τμήματος των εργαζομένων. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν τέτοιε επιχειρήσει που δίνουν μάχη την επιβίωσή του. Οι μόνε που μπορούν να συνεχίσουν να επενδύουν είναι αυτέ που είναι πολύ ισχυρέ οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν να μην ενισχύσουμε αυτέ τι ανισότητε μεταξύ των περιφερειών λόγω των διαφορετικών ικανοτήτων που έχουν οι επιχειρήσει. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά ο κύριος Κάρλο Καλέντα λέει ότι στη φάση της ανασυγκρότησης δεν θα πρέπει να έχουμε διακρίσεις στις επενδύσεις που θα ενισχύουν τις ανισότητες. Και πιστεύω πρώτα απ' όλα θα πρέπει να έχουμε στηρίξη της παραγωγής στην Ευρώπη και διαφύλαξη των θέσεων απασχόλησης. Συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα μπορούσαμε το σχέδιο της ανάκαμψης να το συνδυάσουμε με μια στρατηγική επιστροφή της βιομηχανικής παραγωγής στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η κρίση έχει αγγίξει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες όμως των χωρών μελών θα είναι διαφορετικές ανάλογα με τις διαφορές που έχει η διάρθρωση της οικονομίας τους ή η ανθεκτικότητα των οικονομικών κλάδων ε, στη, στα αποτελέσματα της ε, πανδημίας. Οπότε θα πρέπει τους μηχανισμούς στήριξης να τους προσαρμόσουμε ε, στις ανάγκες και των χωρών της Ευρωζώνης και των χωρών εκτός της Ευρωζώνης. Προτεραιότητα της Ένωσης θα πρέπει να είναι η ανάλογη, αναλογική κατανομή των επενδύσεων μεταξύ των διαφόρων οικονομιών δεν θα πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στο μη CTS του συστήματος εμπορίας εκπομπών, γιατί λιγότερο εύπορες χώρες δεν θα, μερικές φορές καταβάλουν μεγαλύτερη συνεισφορά αντίστοιχα από τις πιο εύπορες και ισχυρές χώρες οικονομικά. Επίσης, ο εισηγητής μιλά για το ρόλο του φυσικού αερίου μεταβατικού καυσίμου Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανάγκη της ασφάλειας των δικτύων και του ανεφοδιασμού σε ενέργεια. Γιατί δεν θα πρέπει να ενδιαφέρομαστε μόνο για το κλίμα, αλλά και για την εξασφάλιση σταθερότητας στην προμήθεια ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις ε, απαραίτητες για μας πρώτες ύλες για την παραγωγή ενέργειας. Σας ευχαριστώ και συγχαρητήρια και ευχαριστώ στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον τελευταίο εισηγητή μας που είναι ο κύριος Μάρκ Μποτεγκά από την ΚΟΕ που αν δεν κάνω λάθος επίσης είναι στην αίθουσα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή μας, τον κύριο Καλέντα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη διαλεκτικότητά του και το πνεύμα συνεργασίας που έχει δείξει με τους και εισηγητές. Ε, ως ΓΚΟΕ φυσικά θα πρέπει να σταθούμε στην κοινωνική και την κλιματική διάσταση. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής. Εγώ εντυπωσιάστηκα κατά τη διάρκεια της κρίσης από από το γεγονός ότι όταν οι εργαζόμενοι είχαν την δυνατότητα να αποφασίσουν, είχαμε αυτοκινητοβιομηχανίες και ε, βιομηχανία αεροναυπηγικής που ε, στράφηκαν στην παραγωγή αναπνευστήρων. Οπότε ε, για μία φορά η βιομηχανία ε, αφουγκράστηκε τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να στραφούμε προς αυτή την κατάσταση για να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως της Σλοβαρδίας που εξάγει όπλα και αναγκάζεται να ε, εισαγάγει ιατροφαρμακευτικό υλικό. Και επίσης με τις δημόσιες επενδύσεις θα πρέπει να εξασφαλίσουμε οι περιφέρειες που σήμερα έχουν πρόβλημα και χαμηλή βιομηχανική δραστηριότητα να μπορούν να αναπτύξουν ε, στο μέλλον διάφορους βιομηχανικούς τομείς με ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Αλλά να μην κάνουμε λάθος στους στόχους. Θα πρέπει να μπει η βιομηχανία στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι η κοινωνία στην υπηρεσία των πολυεθνικών εταιριών. Γιατί είναι κάπως ε, αλλοπρόσελη μια ιδέα που κυκλοφορεί ότι δημιουργώντας ευρωπαϊκά ισοδύναμα ε, της Amazon ή του Lockheed Martin ε, θα εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη κτλ. Αυτό μου φαίνεται επικίνδυνο. Και όταν μιλάτε για Ευρωπαίους πρωταγωνιστές, φοβάμαι μήπως αυτό το πρότυπο έχετε υπόψη. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μια τέτοια στρατηγική θα μετατραπεί σε ένα μαζικό σχέδιο επιδοτήσεων και δωρεάν επιδοτήσεων προς τις πολυεθνικές, που θα μπορούν να παράγουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, επιρρύπτοντας το κόστος των επενδύσεων στην κοινωνία και συνεχίζοντας να καταβάλουν τα ψηλά μερίσματα στους μετόχους τους. Πώς θα πούμε στους απολυθέντες εργαζομένους ότι δεν θα στηρίξουμε αυτούς αλλά στην ουσία τους εργοδότες. Και σήμερα οι πολυεθνικές ε, ζητούν κρατικές ενισχύσεις, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιούνται σε φορολογικούς παραδείσους, συνεχίζουν να καταβάλουν μερίσματα και ετοιμάζονται να προβούν σε απολύσει εργαζομένων. Γι' αυτό είναι παράδεκτο. Και αυτή τη σκέψη θα πρέπει να την συμπεριλάβουμε στη βιομηχανική μας στρατηγική. Θέλουμε ε, ενισχύσεις που θα έχουν κοινωνική ερεσιμότητα και όρους στην εργασία. Επίσης, αξιοπρεπείς θέσεις απασχόλησης ποιοτικέ και ε, επιστροφή της βιομηχανικής και μεταπιτικής παραγωγής στην Ευρώπη. Και θα ήθελα να πω ότι αν η αγορά δεν είναι ικανή να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί ε, να μην αρχίσουμε να δημιουργούμε κάποιους δημόσιους βιομηχανικούς ε, πόλους. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ κύριε Μποτέγκα. Ένα αίτημα έχω μόνο από το KCI ο ε, κύριος Ιγνάσιο Κοράου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω Ιταλικά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ τον εισηγητή για την, το σχέδιο αυτό έκθεσης που αποτελεί μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για να συζητήσουμε πώς θα έχουμε μια νέα αποτελεσματική βιομηχανική στρατηγική. Παραδέχομαι πως ε, θα ήθελα να δω λίγο περισσότερο θάρρος και έμφαση όσον αφορά την πράσινη μετάβαση για την μελλοντική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στο σημείο 15, όπου η έκθεση αφού λέει ότι κάθε κλάδος θα πρέπει να συνεισφέρει στους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρει την ε, σημασία του φυσικού για την ενεργειακή μετάβαση. Ναι, ειδικά όταν μιλάμε για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, χημική βιομηχανία, τσιμέντο, χάλιβα κτλ ε, η οποία αντιπροσωπεύει μόνη της ε, σχεδόν ε, το 14% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε θαραλέοι και φιλόδοξοι ως προς αυτό για να δούμε πώς οι κατασκευαστές αυτών των προϊόντων αλλά και των προϊόντων του αυτοκινήτου θα μπορέσουν να σεβαστούν το περιβάλλον και να έχουμε προϊόντα τα οποία θα φτιάχνονται στην Ευρώπη και θα είναι σωστά. Εύχομαι λοιπόν μετά από όλα αυτά καλή τύχη στον εισηγητή για τις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τον κύριο Μάρκ Νίκλας, ο οποίος είναι τμήματάρχης ε, στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Μας ακούει ο κύριος Νίκλας. Είναι στην αίθουσα ή συνδεδεμένος. Α, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, είχα κάποια προβλήματα σύνδεσης. Να δούμε αν μπορούμε να συνδεθούμε. Εντάξει, θα περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα. Well, if the connection is not uh, I would go to... Αν δεν υπάρχει σύνδεση, πάμε στον κύριο Καλέντα. Και αν ε, ξανασυνδεθεί ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, να του δώσουμε τον λόγο. Για να μην χάνουμε χρόνο. Γιατί έχουμε και τη συζήτηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου θέλουν να μιλήσουν αρκετοί. Δεν έχουμε σύνδεση. Δεν είναι συνδεδεμένο ο κύριος Νίκλας, οπότε μπορείτε να δώσετε τον λόγο. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Καλέντα, έχετε τον λόγο για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας μετά από τις παρεμβάσεις των σκιωδών εισηγητών. Να αναφερθώ σε κάποια από τα σημεία που είπατε. Αυτό το οποίο είπε ο κ. Μπέρεντς είναι ε, σωστό. Πράγματι πρόκειται για χρήματα τα οποία δανειζόμαστε από τις μελλοντικέ ε, γενιές και ακριβώς ε, θα πρέπει να διαχειριστεί η Κομισιόν τα χρήματα αυτά με τρόπο ώστε να ωφεληθούν και οι μελλοντικέ γενιές από μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Μετά ο συνάδελφος είπε κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν ε, είχα πει. Έχουμε την σημασία των ε, δημοσίων προμηθειών, η οποία τονίζεται αφενός στην έκθεση και η σημασία του να ξαναδούμε την στρατηγική για τον ανταγωνισμό της νομοθεσίας αντιτράστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πω πως ε, όσον αφορά τις Ευρωπαίους πρωταθλητές, πως κατά κανόνα πληρώνουν καλύτερα τους εργαζόμενους τους. Αλλά εμείς έχουμε μια έκθεση η οποία ακριβώς έχει στόχο να προσθετεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις ε, μεγάλες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται καλύτερη επίβλεψη. Επίσης αναφέρθηκε πολλές φορές η σημασία του Just Transition Fund και του κοινωνικού μετασχηματισμού και προστασίας και όπως ξέρετε ότι όταν λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένους ε, τομείς όπως ο τουρισμός ε, και η μηχανία, όπου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία τώρα. Για το θέμα του φυσικού αερίου ο ή αναφέρθηκε αφενός στο χάλιβα φετερού στο φυσικό αέριο. Ο μοναδικός τρόπος για να μην έχουμε άνθρακα στο ε, χάλιβα είναι το φυσικό αέριο. Για να αντιληφθούμε λοιπόν την δυσκολία στην έκθεση αυτή, το παράδειγμα του χάλιβα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί εάν θέλουμε να μην υπάρχει χάλιβα στην παραγωγή πρέπει πρώτον να χρηματοδοτήσουμε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό. Οπότε νέα εργοστάσια. Δεύτερον, να υπάρχει ένας μηχανισμός αντιστάθμισης άνθρακα, κάτι το οποίο αναφέρθηκε χθε από την Κομισιόν. Τρία, να υπάρξει μια ε, επιδότηση του φυσικού αερίου, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική πηγή ενέργειας για την παραγωγή χάλιβα. Οπότε είναι μια μεταβατική ε, ενέργεια, το φυσικό αέριο, οπότε πρέπει να επιλέγουμε πάντα ε, μεταξύ φυσικού αερίου και ε, άνθρακα, οπότε νομίζω αξίζει τον κόπο να επιλέξουμε το φυσικό αέριο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, να σας υπενθυμίσω ότι η παρθεσμία για τις τροπολογίες είναι Δευτέρα 22 Ιουνίου. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμα και παρακαλώ. Σας παρακαλώ να καταθέτε στο μέτρο του δυνατού στα αγγλικά και να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κύριο Καλέντα, ευχαριστώ τους Διερμηνείς. Περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη σχετική πολιτική. Όπως ξέρετε, η ΙΤΡΕ έχει ζητήσει την άδεια για μια εκθέση ιδίας πρωτοβουλίας. Ε, δεν έχει εγκριθεί ακόμα από την διάσκεψη των Προέδρων. Ο κ. Ε, Παύλο Μπορκία, ξενόματος ομάδας ID, είναι ο εισηγητής, υπεύθυνος για αυτή την έκθεση. Η έκθεση όμως δεν έχει ακόμα εγκριθεί, οπότε σήμερα θα γίνει μια γενική έτσι, ανταλλαγή απόψεων για την πολιτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δεν θα συζητήσουμε την έκθεση. Έχουμε τον ίδιο χρόνο, 35 λεπτά. Βεβαίω, για πού μιλάμε για τέλος για απόψεις; Έχουμε έναν κατάλογο πολιτών, τόνο που μιλάμε για ανταλλαγή απόψεων, έχουμε έναν κατάλογο μιλτών, τον οποίο έχουμε ήδη συζητήσει με τις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στους ε, συναδέλφους ε, και ο πρώτος στον κατάλογο των ομιλητών είναι ο κύριος Έλερ, εξ του ΕΛΚ. Um, so... Τώρα είμαστε σε μια περίεργη συζήτηση κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε πρόταση για να συζητήσουμε. Ήδη το Μάρτιο ε, ε, έχει οριστεί αυτή η ημερήσια διάταξη από την ε, Κομισιόν. Για τις μικρομεσαίες ανησυχώ πραγματικά, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά το σχέδιο ανάκαμψης, το χτεσινό, χθες το βράδυ πήραμε τις λεπτομέρειες, δεν γίνεται αναφορά στις μικρομεσαίες και αυτό είναι πολύ, πολύ προβληματικό. για ανησυχώ Γιατί όταν κάνει προτάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει αυτέ να είναι συνεκτικές. Δεν μπορεί να πηγαίνουν προ πάσα κατεύθυνση. Ανακοινώσανε ότι θέλουν να κάνουν κάτι για τις μικρομεσαίες, από την άλλη μιλάμε για το κλιματικό νομοσχέδιο και την ε, βιομηχανική πολιτική. Όλα αυτά πώς συνάδουν, πώς συνδέονται μεταξύ τους και τι γίνεται με τις μικρομεσαίες που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν δείτε ε, το ιστορικό ε, του θεματολογίου για τη βιομηχανική πολιτική, Καμία ε, βιομηχανική πολιτική δεν επέτυχε, ούτε είχε ισχυρή ε, στόχευση στις μικρομεσαίες και τώρα στο σχέδιο ανάκαμψης το αφήνουν πλήρως στα χέρια των κρατών μελών να δουν τι θα κάνουν με τις μικρομεσαίες και σε ποιο βαθμό. Αν δούμε τα χρηματοδοτικά μέσα, δόθηκε σκληρή μάχη για να υπάρξει ειδικό εργαλείο μέσα σε αυτά τα ε, χρηματοδοτικά για τις μικρομεσαίες, για τη γενοτομία και γενικότερα θα προσπαθήσουμε αυτό κάπως να το περιορίσουμε και προσπαθήσαμε, αλλά είναι ανησυχητικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Στο πρόγραμμα Horizon ε, έχουν κάνει περικοπές στην Ιταλία, στην Ισπανία, στα προγράμματα των μικρομεσαίων. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να μην το πληρώσουν οι μικρομεσαίες και να μην είναι κενά λόγια αυτά που ακούμε και ακούφια για τις μικρομεσαίες. Χρειαζόμαστε πιο πολλές συνεκτικές πολιτικές ε, πριν αρχίζουμε να χαράσουμε διάφορες στρατηγικές για τις μικρομεσαίες, για το κλίμα, ε, για ε, τη βιομηχανία. Τι συγκεκριμένη η κλιματική νομοθεσία. Ε, είναι δυνατότητα για τις μικρομεσαίες και ευκαιρία, αλλά είναι και απειλή. Είναι πολύ γενικόλογα και αόριστα αυτά. Από τη σκοπιά του ΕΛΚ, λοιπόν, βεβαίως και θα πρέπει να θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι προτεραιότητα και τομέα που μας ανησυχεί αλλά που έχει και δυνατότητες στην Ευρώπη. Αλλά δεν έχει νόημα να έχουμε έτσι κατακαιρματισμένες πολιτικές, ασύνδετες μεταξύ τους. Και το προηγούμενο θύμα, μια μάλλον το πρώτο θύμα μια τέτοια ε, κατάστασης είναι οι μικρομεσαίες. Γιατί η μηχανία θα βρει το δρόμο της και τη χρηματοδότησή της και θα τα πάρει είναι οργανωμένοι, ε, είναι έμπειροι, ξέρουν πώς να ζητούν τις ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, πώς να κάνουν τις αιτήσει. Η στρατηγική για τις μικρομεσαίες είναι πάρα πολύ κρίσιμη και για το κλίμα και για τη βιομηχανική πολιτική και για το σχέδιο ανάκαμψης. Και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν κοιτάμε μια πρόταση απλώς του Μαρτίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει αυτό να είναι ένα εγκάρσιο θέμα που να διαπερνά όλες τις προτάσεις που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη και την Πράσινη Συμφωνία και ακόμα περισσότερο με κάτι που μου λείπει από εδώ να γίνεται η ίδια προσπάθεια για το σχέδιο ανάκαμψης ε, και για μια ψηφιακή ανάκαμψη. Γιατί αυτό είναι το κλειδί για την, ε, ε, τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες, οι οποίες υπολείπονται. Οι μεγάλες βιομηχανίες μπορούν εκεί να επενδύσουν και στα ψηφιακά, οι μικρομεσαίες την πληρώνουν. Ευχαριστώ πολύ για τον πρώτο γύρο Έχουμε τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, δύο λεπτά και στο δεύτερο γύρο ένα λεπτό. Παρακαλώ να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα. διάγραμμα. σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Κουταχάρ. Γεια σας. ακούτε? Ναι, ναι, σας ακούμε. Και σας βλέπουμε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε η συζήτηση αυτή που αρχίζει σήμερα για τις μικρομεσαίες είναι πολύ διαφορετική από αυτή που θα είχα φανταστεί πριν από λίγους μήνες. Πάντως θα πρέπει να θυμηθούμε πόσο ε, ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός εξαρτάται από τις μικρομεσαίες. Πολλές είναι και οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Υπηρεσίες, τουρισμός, κατασκευές. Ε, είναι λίγοι από τους τομείς μόνο των μικρομεσαίων. Πραγματικά είναι η ραχοκοκαλιά του παραγωγικού μας συστήματος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε αρχές Μαρτίου μία ανακοίνωση που έχει πολλές και πολύτιμες προτάσεις, αλλά φυσικά δεν περιλαμβάνει το COVID που έχει τώρα επιπτώσει σε όλες τις μικρομεσαίες και στους εργαζομένους και στην ε, θέση τους στην αλυσίδα παραγωγής και στις αγωνίες που αντιμετωπίζουν θα πρέπει οπωσδήποτε όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη τους επόμενους μήνες και να συζητήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τις προτεραιότητες ε, της δίκαιης, της σωστής μετάβασης, να προσαρμοστούμε στη νέα φάση. Το COVID-19 έχει συμπαρασύρει πολλές βεβαιότητες. Αλλά το ψηφιακό χάσμα των μικρομεσαίων και η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής παραμένουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές εταιρείες μας να γίνουν πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές παγκόσμια. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στην κυρία Μαρτίνα Ντλαμπαϊωβά από τη Ρινιού. Παρακαλώ. Hello, can you, can you hear me? Αγαπητοί συνάδελφοι, πολύ χρήσιμη και η τωρινή συζήτηση και η προηγούμενη και πολύ επικοδομητικές. Νομίζω ότι είναι κρίσιμο να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά για να εξασφαλίσουμε μια συνέργεια μεταξύ τη ε, βιομηχανική στρατηγική και τη στρατηγική για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και αυτό προ όφελο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το διακύβευμα είναι εκατομμύρια θέσει απασχόληση Και θα πρέπει να συνδυάσουμε όλα τα μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μα για να εξασφαλίσουμε ανάκαμψη. Βέβαια, ο διάβολο βρίσκεται στι λεπτομέρειε. Θα πρέπει να αναλύσουμε τις συγκεκριμένες επιπτώσεις που θα επιφέρει το σχέδιο ανάκαμψης στο οικονομικό τοπίο και να δούμε όχι μόνο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, δύο-τριών επόμενων χρόνων, αλλά και μέσω πρόθεσμα μέσα στην ευθετία. Και ο σκάδιμος μας ηγητής σε αυτό και το θέμα της ε, βιομηχανικής στρατηγικής ε, είναι ε, υπέρ της επίλυση του προβλήματος της ρευστότητας, ε, της έλλειψης ρευστότητας και επίσης ε, να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προβούν σε αυτό το ψηφιακό ε, μετασχηματισμό και να εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ισότιμες ευκαιρίες σε όλες τις χώρες μέλη, ανεξάρτητα που έχουν την έδρα τους λοιπόν οι επιχειρήσεις. Επίσης, έχουμε και κάποιες προτεραιότητες που στο ισχυόν πλαίσιο είναι ακόμη πιο σημαντικές. Θα σταθώ σε δύο. Καταρχήν, οριζόντιος στόχος ε, πλούστευσης ε, και ε, του εφνομοθετήν. Επίσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται ισότιμα στις μικρομεσαίες οποιαδήποτε νέα πρόταση και η πρόταση run in και run out. Επίσης, όσο θα αναλύσουμε τα, κράτη, τα μέσα που έχουν τα κράτη-μέλη, θα πρέπει όλα να συνειδητοποιήσουν ότι θα πρέπει να εξορθολογήσουν τις δράσεις τους και να είναι αυτόματη αρχή η αρχή της, του ψηφιακού μετασχηματισμού. Θέλουμε ανθεκτικά βιομηχανικά συστήματα και αυτό το καταφέρουμε μόνο με ισχυρή συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και να του δώσουμε ευκαιρία για να επιβιώσουν από την κρίση και να του προστατεύσουμε από αφαιρέγγιου οφειλέτε, είτε είναι επιχειρήσει είτε είναι το κράτο. Συμφωνώ με τον κύριο Έλερ για το Ταμείο Ανάκαμψη. Χθε βράδυ αναζητούσε συγκεκριμένες μνήες ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δεν βρήκα τέτοιες συγκεκριμένες μνήες. Οπότε είναι σημαντικό ε, να είμαστε εισπυρωμένοι ως μέλη και ως Επιτροπή της Ήτρε στα θέματα αυτά και προσβλέπω σε στενή συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ομάδα ID. Ο κύριος Πάολο Μπόρκια που είναι και ο εισηγητή τη έκθεση εφόσον δοθεί άδεια για τη σύνταξη τη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα τα Ιταλικά. Πρώτα απ' όλα, εν αναμονή της ε, έγκρισης ε, της έκθεσης θα πρέπει οπωσδήποτε να καθυστερήσουμε λίγο για να ξεκινήσουμε μετά να εργαζόμαστε στην έκθεση για να δούμε ακριβώς πρώτα απ' όλα και τι επίδραση θα έχει η επιδημία. Όμως θεωρώ, έχοντας ως αφετηρία την ανακοίνωση της Κομισιόν της 10ης Μαρτίου, να φτάσουμε σε μια διόρθωση, όπως ακριβώς είπε η κυρία Κουταγιάρ. 10 Μαρτίου είχαμε την έκθεση, 11 Μαρτίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προκήρυξε πανδημία. Όμω για τι παρεμβάσει των συναδέλφων. Εγώ συμφωνώ πλήρω με τις ανησυχίε ε, των συναδέλφων Έλερ και Χλαμπάιοβα, ε, αυτό δηλαδή το οποίο είπαν ε, για αυτό το, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίε επιχειρήσεις και τα όσα ανέφερε χθε στην Ολομέλεια η κυρία Φόντερ Λάιεν. Βεβαίω η ανάκαμψη θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις γιατί ε, αυτή τη στιγμή είναι στα όρια της χρεοκοπίας κάποιοι ε, κλάδοι αντιμετωπίζουν κρίση ανεπανάληπτη. Αυτό φαίνεται ούτως ή άλλως από τους αριθμούς. Θεωρώ λοιπόν πως η στρατηγική αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αποτελέσει ένα συγκεκριμένο και αποτελεσματικό μέσο το οποίο θα στηρίζεται από επαρκείς ε, πόρους ε, που θα κατευθυνθούν ακριβώς εκεί πέρα που υπάρχει το πρόβλημα γιατί το κείμενο αυτό βεβαίως θα πρέπει να είναι συνολικό, τεχνικό και κυρίως ρεαλιστικό έτσι. Να μην αναφερόμαστε σε άλλες ε, προηγούμενες ε, καταστάσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναφερθούμε πολύ συγκεκριμένα σε διάφορα θέματα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ε, των μικρομισίων επιχειρήσεων. Η πραγματικότητα της υποκεφαλαιοποίησης του κόστους της γραφειοκρατίας, το οποίο είναι δυσανάλογο σε κάποια κράτη ε, σε σχέση με άλλα. Να δούμε επίσης το θέμα της καθυστέρησης των πληρωμών, της διαφοράς, ε, της παραγωγικότητας μεταξύ των χωρών, αλλά επίσης και του θέματος ε, των στρεβλώσεων αλλά και το τι μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Επίσης υπάρχουν άλλα θέματα όπως οι φόροι για τον άνθρακα στα εξωτερικά σύνορα ε, που θα κάνουν νομίζω το κείμενο ακόμη πιο πλήρες σε σχέση με αυτό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή. Σας, Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Ένερη Χάν. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, 20 εκατομμύρια ε, στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ε, τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Και μάλιστα οι περισσότερες, 90% των επιχειρήσεων λένε ότι έχουν χάσει τους πελάτες τους και γι' αυτό θα πρέπει τη χρηματοδότηση να την κάνουμε προσβάσιμη στις μικρομεσαίε επιχειρήσεις. Χθε ακούσαμε το νέο σχέδιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση τη Νέα Γενιά, προκειμένου να δοθεί στήριξη φερεγγιότητας στις μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει τη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από τα υπάρχοντα προγράμματα. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη ευκαιρία να, ε, να χρηματοδοτήσουμε και την οικολογικό μετασχηματισμό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητά τους για να στραφούν προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, αξιοποιώντας και τα κονδύλια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης. Μην ξεχνάτε και την πράσινη συμφωνία που θα δώσει ευκαιρίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό δεν το τονίσαμε επαρκώ στην στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Μαρτίου. Θα πρέπει να το βελτιώσουμε και θέλουμε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και γι' αυτό η βιομηχανική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να έχει ειδικά εργαλεία για να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να τις ενημερώσει για τις ε, πράσινες ευκαιρίες που έχουν και τα φιλοπεριβαλλοντικά και οικολογικά εργαλεία. Έχουμε μια μονοδική ευκαιρία να χωράξουμε τον κόσμο, το δρόμο για μια βιώσιμη ε, οικολογική ε, οικονομία στην Ευρώπη. Χάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά και στον ε, περιβαλλοντικό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Ευχαριστώ. ECR. E το λόγο έχει ο κύριος από το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα σοφά λόγια του συναδέλφου από το ΕΛΚ του κυρίου Έλλερ με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να λάβω μέρος στη συζήτηση, αν και δεν έχω μεγάλη πείρα με το ενωσιακό δίκαιο, ούτε είμαι τόσο εξοικειωμένος όπως άλλοι προλαλήσαντες, αλλά για 20 χρόνια ήμουν επιχειρηματίας και έχω πολύ πλούσια πείρα, γιατί είδα το ενωσιακό δίκαιο στην πράξη. Και σίγουρα ο επιχειρηματίας αγαπά τα προϊόντα που παράγει και πουλάει, αλλά ε, αναλαμβάνει και πολλούς κινδύνους, ε, γιατί δεν είναι απλώς ένας διαχειριστής επιχείρησης. Όταν μια εταιρεία φτωχεύει, μπορεί ο επιχειρηματίας να χάσει τα πάντα. Και αν οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να λένε ότι θα πρέπει να τηρήσετε νέους κανονισμούς και νέες διατάξεις, μερικές φορές ε, ε, ε λέμε ότι δεν αξίζει όλη η προσπάθεια. Και μάλιστα με τον ε, Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων ε, χρειάστηκε να πουλήσω όλες μου τις εταιρείε. γιατί ε, είχα την αίσθηση ότι είχα πόλεμο με την κάθε κυβέρνηση και με το ε, ενωσιακό δίκαιο και σίγουρα ο κανονισμός GDPR με κατέστρεψε. Και τώρα έχουμε την κρίση που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στι επιχειρήσει. Πολλοί μίλησαν για ευκαιρίε εδώ, αλλά μόνο για του επίλεκτου λίγου. 95% των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή ε, πασχίζουν για να επιβιώσουν. Οπότε θα πρέπει να, για να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μειώσουμε πρώτα την ομοθεσία, να την απλουστεύσουμε και αν θέλουμε ε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον θα πρέπει να επενδύσουμε στην καινοτομία. Πρώτα καινοτομία και μετά ε, νομοθετική ρύθμιση. Επίσης, θα πρέπει να διδαχθούμε από τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε και το Ισραήλ. Εκεί ε, η αμυντική βιομηχανία είναι καλός πελάτης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από εκεί, από αυτές ξεκινάει η καινοτομία. Και εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να μιμηθούμε αυτές τις χώρες και με τη βιομηχανία του διαστήματος. Επίση, χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το καθήκον φροντίδα των τραπεζών είναι τόσο μεγάλο γιατί ε, οι διατάξεις από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 δυσκόλεψαν τα πράγματα και τελικά οι τράπεζες δεν είναι λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να, γεφυρώσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο με τις ε, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζονται οικονομικό σύμβουλο και όχι σύμβουλο βιωσιμότητας. Ας κάνουμε αυτή τη γέφυρα. Ο κύριος Ποτεγκά επίσης είναι στην αίθουσα και θα μας μιλήσει εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Πρώτον, ε, συμφωνώ. Ε, δεν καταλαβαίνω καθόλου απολύτως γιατί έχουν ξεχάσει ε, ε, ε χτες το σχέδιο ανάκαμψης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πολύ λυπηρό αυτό, πολύ δε περισσότερο που απέναντι στην κρίση δεν είναι ίσες όλες οι επιχειρήσεις. Υποφέρουν πολλές μικρομεσαίες, ενώ κάποιες μεγάλες ηλεκτρονικού εμπορίου, ε, διανομής, ε, Amazon, Carrefour, Colruyt στο Βέλγιο, ε, αυξάνουν τον τζίρο τους και μέχρι και 20% αυτό που θα ήταν χρήσιμο κατά τη γνώμη μου είναι να δούμε πώς μπορούμε να ε, οργανώσουμε ε, μία μεταφορά αλληλεγγύης από αυτές τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές, τις διανομής που έχουν αυξήσει τα κέρδη τους προς τις μικρομεσαίες που δυσκολεύονται. Ένα αυτό. Δεύτερο, πιστεύω ότι υπάρχουν και ιστορικά παραδείγματα στις ε, Ηνωμένε Πολιτείε, μετά τον πόλεμο θα μπορούσε να είναι και αυτή μια ιδέα ε, φορολόγησαν τα υπερκέρδη. Θα μπορούσαμε να τα φορολογήσουμε κατά 75% και πώς ορίζονται τα υπερκέρδη ανάλογα με τα κέρδη του ίδιου μήνα σε προηγούμενα έτη. Επίσης θα πρέπει να εγκαταλείψουμε οποιαδήποτε απόπειρα διεύρυνσης ε, ε του, ε, των κριτηρίων και των ορισμών ε, μικρομεσαία επιχείρηση είναι αρκετά ε, ευρύς ο ορισμός στην Ευρώπη της μικρομεσαίας επιχείρησης για να δίνονται χρήματα σε επιχειρήσεις που δεν είναι τόσο μικρές ούτε πολύ μικρές. Ε, και τέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, ξαναδούμε τις εταιρείε μεσαίας κεφαλαιοποίησης προς τα κάτω με αρνητικό τρόπο αυτά τα mid-cap. Αυτός είναι ένας τρόπος να δίνουν λεφτά σε εταιρείε που είναι κανονικές επιχειρήσεις. Αλλά είναι πολύ μεγάλες για να είναι μικρό μεσαίες, ε, οπότε ας αναλάβουν τις ευθύνε τους. Δεν κατάλαβα τι τις χαρακτηρίζουμε mid-cap και τις βοηθούμε όλες με τον ίδιο τρόπο. Έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα ε, ε μεγαλύτερες και χάνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα που θα είχαν οι μικρότερες, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποτέγκα. Περνάμε στο δεύτερο γύρο των μελών της ΣΥΤΡΕ, όχι εξ ονόματο των πολιτικών τους ομάδων, τα μεμονωμένα μέλη, αλλά τώρα έχετε ένα χρόνο έκαστο. Το πολύ. Για να προλάβουμε να τελειώσουμε γέρο. Αρχίζω λοιπόν με την κυρία Βίρκουνεν. Ναι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας συνάδελφοι. Νομίζω ότι ακούστηκαν πολλά ωραία. Επίσης, οι μικρομεσαίες είναι πραγματικά η αχοκοκαλιά της οικονομίας και φυσικά θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτές. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που έχουν βγει από αυτό το κεφάλαιο που είναι πολύ μικρές και μπορεί να είναι μεσαίας κεφαλαιοποίησης αλλά δεν είναι μεγάλες μπορεί να είναι πολύ μικρές. Ακόμα και οικογενειακές. Και θα πρέπει να τις φροντίσουμε και αυτές, διότι αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις και δυσκολίες. Γενικά όμως το σημαντικότερο είναι να ασχολούμαστε με τη χρηματοδότησή τους και την άντληση κεφαλαίων. Ε, θα πρέπει όπως ακούσαμε και προηγουμένως, να ε, έχουμε ένα πλαίσιο καινοτόμο, κανονιστικό για να κοιτούμε εναλλακτικέ μορφές ενίσχυσης. Γιατί και οι ίδιε επιχειρήσεις είναι πηγές καινοτομία και μπορούν να μας βοηθήσουν με την ψηφιοποίηση κτλ. Είναι πραγματικά, επαναλαμβάνω, η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μας και αξίζει να εστιάσουμε σε αυτές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βίρκουνεν. Η κυρία Τόγια, παρακαλώ, αντιπρόεδρος μας. Can I speak? Yes, we can hear you, but not okay. the camera is not well uh, adjusted at your face. Grazie. Eh, vorrei innanzitutto, vorrei innanzitutto... Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα... Α. Toia potrebbe cambiare la... la... Αλλάξτε την κάμερα.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 Πατήστε το κουμπάκι που δείχνει μια κάμερα. Ναι, το έκανα, το έκανα. Αλλά δεν δουλεύει. Θα ανανεώσουμε την σελίδα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα επανέλθουμε στην κυρία Τόγια. Ας ακούσουμε την κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ε, εν τω μεταξύ η γραμματεία έρθει σε επαφή με την κυρία Τόγια να τη βοηθήσει λίγο. Και θα επανέλθουμε όταν είναι έτοιμη. Τον λόγο έχει η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Buenos días. Καλημέρα σας και ευχαριστώ. Θα ήθελα πραγματικά να ενθαρρύνω και εγώ να αναγνωρίσουμε περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, που είναι πραγματικά η ραχοκοκαλιά. Ε, δεν θα πρέπει να είναι σε μειονεκτική θέση. Οι μεγάλες εταιρείες έχουν φορολογικά ε, κίνητρα, ελαφρύνσεις, ρευστότητα ε, και δυνατότητα δανεισμού. Οι μικρομεσαίες όχι. Χρειαζόμαστε ειδική γραμμή χρηματοδότησης αποκεντρωμένη που να είναι κοντά ε, στους επιχειρηματίες και ε, στον τόπο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Για να είναι καλύτερη επίσης και η επαγγελματική εκπαίδευση και εκπαίδευση γενικότερα να μην υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία της εκπαίδευσης με τις ε, δεξιότητες που ζητούν οι εταιρείε. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει ένα μειογενές πρόγραμμα στην Ευρώπη ε, και ελπίζω εδώ να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική υπέρ της επιχείρησης χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι βελτιώνεται καλύτερα όλο το πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων. Ενέργεια. Ε, πρέπει επίσης να τη λάβουμε υπόψη σε πλαίσια της εφορίας και της πράσινης οικονομίας και του Πράσινου Συμφώνου. Τώρα θα πάμε στην κυρία Αγγέλικα Νίμπλερ. Έχετε το λόγο. Γεια σας. Εδώ, ε, Αγγέλικα Νίμπλερ, ευχαριστώ πολύ, ε, Πρόεδρε. Έχω ένα λεπτό μόνο είναι πολύ σημαντικά τα θέματα, αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, ότι ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις βάζουμε σε όλα μας τα πολιτικά προγράμματα και σε όλες τις πολιτικές μας. Μελέτη αντικτύπου, τεστ για τις μικρομεσαίες, όχι νέα θέματα, θα δεν είναι καινούργια αυτά, πρέπει να τα θυμόμαστε όλα. Όλα αυτά που προτείνονται ε, και στα πλαίσια του πακέτου ανάκαμψης, τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι θα πρέπει να διορθώσουμε, να αναπροσαρμόσουμε ε, πάντα σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ένα δεύτερο θέμα, μείωση της γραφειοκρατίας. Πάρα πολύ σημαντικό να μην έχουν άσκοπες επιβαρύνσεις διοικητικές ε, διαφορές υποχρεώσεις ενημέρωσης, τεκμηρίωσης και πάει λέγοντας που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη λειτουργία τους. Ό,τι μπορούμε να ε, ελαφρύνουμε εκεί θα είναι κέρδος. Ή τα διάφορα αυτά υποχρεωτικά που επιβάλλουμε στις επιχειρήσεις, καλό είναι να τα αφήσουμε στην άκρη για κάποιο διάστημα μέχρι να περάσουν αυτό το γκάβο. για να δούμε τι συγκεκριμένα σημαίνουν όλα αυτά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Danke. I go now to Mr. Ευχαριστώ. Θα περάσω τώρα στον κύριο Χάισεν. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κρίστια. Συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που μας είπαν ότι οι μικρομεσαίες αξίζουν καλύτερη θέση ε, σε όλη τη στρατηγική ανάκαμψης ε, και καταπολέμησης των απολειών ε, και του κόστους που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός. Αν θέλουμε πραγματικά η οικονομία μας να ανακάμψει και να ζήσουν οι μικρομεσαίες, θα πρέπει και να τις υποστηρίξουμε για να περάσουν αυτό το μετασχηματισμό που χρειάζεται και να ε, ε, υπερκεράσουν τα εμπόδια. και όλες αυτές τις ανητικές επιπτώσεις κοινωνικές και οικονομικές της κρίσης του κορονοϊού. Από την άλλη, Είναι πολύ καλό αυτό για μένα ως ε, εισηγητή για το Ταμείο δίκαιη μετάβαση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει συνδέσει. Αυτό σαφέστατα. Γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το, ανήκουν, το αξίζουν συγγνώμη, και θα πρέπει να τις βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. We go back now to... Ευχαριστώ. Κύριε. Ευχαριστώ. Ε, θα γυρίσουμε τώρα στην κυρία Τόγια που νομίζω έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. It's okay now. No. Not really, but please proceed, Patricia. Please. Uh, ε, Πατρίσια, μπορείτε να πάρετε το λόγο. Η κάμερα δεν έχει τελείως αποκατασταθεί, αλλά δεν πειράζει. No. Uh, Madame Toya, we can... No. Not my the...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 Θέλω μόνο να συμφωνήσω με την ανησυχία που εξέφρασαν όλοι οι συνάδελφοι, η οποία δείχνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, χάνονται από το ραντάρ της ευρωπαϊκής πολιτικής. Είναι λοιπόν ο δικός μας ο ρόλος εδώ σε αυτή την Επιτροπή να τους επαναφέρουμε στο επίκεντρο της ε, προσοχής με συγκεκριμένες ε, πράξεις. Τα προβλήματα είναι ξεκάθαρα πρόσβαση στην πίστοση, πρόβλημα ε, ρευστότητας ε, και τεχνολογίες ε, Ακριβώς ο μετασχηματισμός ο τεχνολογικός και ο περιβαλλοντικός θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε μια ανάλυση των προβλημάτων τους. Αλλά κάτι συγκεκριμένο είναι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει γιατί μειώνεται ο προϋπολογισμός για το κόσμο, για την έρευνα και την καινοτομία Οπότε θα πρέπει να γίνει κάτι και όσον αφορά τους όρους χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε τώρα στον κύριο Μπεντλάγκη από τους Πράσινους. Κύριο Προφανώς ε, καλωσορίζουμε αυτό το πρόγραμμα, αλλά είναι γεγονός ότι δεν επαρκεί και δεν αναφέρεται αρκετά η πτυχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, ε, ανησυχητικό για εμάς είναι ότι στο παρελθόν, το μιλούσαμε για Ευρωπαίους πρωταθλητές, ε, ήταν διαφορετικό το αφήγημα τώρα, ας πούμε, λέμε ότι πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας. Εμείς όμως θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα Πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε ότι σε όλα τα προγράμματα θα επανέλθουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο. Δεύτερον, να έχουμε ειδικά κονδυλία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να γίνει ο ψηφιακό μετασχηματισμός και ο οικολογικός μετασχηματισμός που απαιτείται αλλά επίσης να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε δίκαιη πρόσβαση όλων στις αγορές ε, για να υπάρξει ακριβώς ε, ανθεκτικότητα στις μικρομεσαίε επιχειρήσει, να μην εστιάζουμε σε μεγάλους Ευρωπαίου πρωταθλητές. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Πιλάρ Ευχαριστώ κύριε Μποσελάγκερ. Η κυρία Πιλάρ τώρα. Tiene la palabra. Έχετε το λόγο, κυρία Δελκαστήγιο. Συμφωνώ με πολλούς προλαλήσαντες που με κάλυψαν αρκετά. Δυστυχώς ο ήχος είναι πάρα πολύ κακός από την κυρία Πιλάρ principle need to be an integral part of the youth recovery plan. More specifically, it's paramount that the recovery plan helps channel our SME strategy, providing SMEs with adequate human resources as well as... Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να γίνουν πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές στην οικονομία όπως έχει μεταμορφωθεί. Αλλά η ψηφιοποίηση είναι πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτή. Και σίγουρα οι χθεσινές προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες από πολιτική άποψη, αλλά υπάρχει μεγάλη ανισορροπία μεταξύ του περιβαλλοντικού πυλώνα και του ψηφιακού πυλώνα της πρότασης. Όχι μόνο ως προς τη χρηματοδότησή τους, θα πρέπει να καλύψουμε το επενδυτικό χάσμα που υπάρχει, που είναι 120 δις σε σχέση με, το περιβαλλοντικό, με την περιβαλλοντική χρηματοδότηση. Υπάρχει 120 δις επενδυτικό χάσμα μεταξύ ψηφιακού πυλώνα και περιβαλλοντικού πυλώνα και θα πρέπει να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα. Έχουμε ευθύνη ως μέλη της Επιτροπής Ήτρε να μεριμνήσουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κάλυψη αυτού του χάσματος γιατί είναι σημαντική η ψηφιοποίηση και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πιλάρ. Τελευταίος μιλητή στον κατάλογό μας, ο κύριος Πιέτρο Φιόκη. Μην ξεχνούμε και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα με τον ορισμό. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι ο αδύναμος κρίκος αυτής της οικονομικής κρίσης. Πρώτον, γιατί έχουν πληγεί και από τον κανονιστικό αντίκτυπο της Νέας Πράσινης Συμφωνίας αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και δεν έχουν ούτε τη δομή ούτε τους πόρους να προσαρμοστούν και επίσης έχουν πολύ περισσότερα προβλήματα από τις μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις στην ε, πρόσβασή τους ε, στα κοινοτικά κονδύλια, κυρίως για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Οπότε θα ήθελα να τονίσω τη σημασία που έχουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι μικροσκοπικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Μόνο στην Ιταλία είναι το 65% ε, το, το, αλλά και στην, Ιταλ... στην Ελλάδα, στην Ισπανία, την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος των πολύ μικρών επιχειρήσεων ε, και η συμμετοχή τους στο Εθνικό ΑΕΠ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φιώκη. Έχουμε και προσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ σημαντικό, γιατί καμία στρατηγική δεν νοείται χωρίς ε, καλό συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστούν σωστά οι πολιτικές. Έχουμε την κυρία Κριστίν Σράιβερ, που είναι διευθύντρια στην ε, Γενική Διεύθυνση Grow, αλλά και την κυρία Μάριτ Νάιμαν, που είναι αναπληρώτρια τμήματάρχη στην ίδια Γενική Διεύθυνση, τη Γενική Διεύθυνση Grow τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οπότε θα δώσω το λόγο για σύντομε παρεμβάσει στην κυρία Σράιβερ. Χωρίς μικρόφωνο, δυστυχώς, η ομιλήτρια. Ε, il faudra appuyer sur le bouton ε, speak. Ε, excuse me, I have also two interventions from, from... Έχω δύο παρεμβάσεις από το ΚΑΤΣΤΙΑΕ. Επειδή βλέπω ότι φεύγει ο κύριος Μπελαμή, ε, να ακούσουμε πρώτα την κυρία Σράιμπερ και μετά... Ή μάλλον όχι, οι συνάδελφοι που ζήτησαν το λόγο. Α, κυρία Σράιμπερ, θα σας δώσω το λόγο, αλλά προηγουμένως ο κύριος Μπελαμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ε, όλοι αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν στο σχέδιο ανάκαμψης που μας παρουσιάστηκε χθε να ξεχάσαμε κυριολεκτικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μα είναι το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Πάνω από 60% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς είναι εκείνε οι εταιρείε οι οποίες βρίσκονται πιο εκτεθειμένες τώρα στην κρίση του κορονοϊού και οι επιχειρηματίες οι ίδιοι αυτοί πρέπει να πάρουν τα μεγαλύτερα ρίσκα και χωρίς καμιά αμφιβολία είναι και στην πιο εύθραυση κατάσταση σήμερα και φυσικά θα πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο οποιασδήποτε ε, μορφής σχεδίου ανάκαμψης, ιδιαίτερα αν αυτό είναι δάνειο. Από την αρχή της συζήτησης αυτής μιλάμε για ποσά που θα δαπανίσουμε, αντί να συζητάμε ε, για το πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Εάν ε, δανειστούμε, που προσωπικά πιστεύω ότι είναι μεγάλο ρίσκο, θα πρέπει να το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, ώστε αύριο οι μελλοντικέ γενιές που θα κληθούν να αποπληρώσουν το δάνειο αυτό, να έχουν την οικονομική δυνατότητα να απομισθούν αυτό το βάρος. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να εγγυηθούμε ε, την ευημερία τους και άρα να έχουν αντέξει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπελαμή για την παρουσία σας. Η κυρία Τελαπίσα Καριών, ένα λεπτό το πολύ. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή να δούμε την ανθρώπινη διάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, συχνά φαίνεται να έχουμε στο μυαλό μας μεγάλους οργανισμούς, ε, ε, ογκώδεις. Μα μικρομεσαία επιχειρήση μπορεί να είναι και ατομική, δύο ατόμων ή οικογενειακή, που έχουν τεράστιες ε, προκλήσεις να αντιμετωπίσουν, χρέη, ε, και δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πολλές φορές έχουν υποθηκεύσει τα σπίτια τους, έχουν βάλει περιουσιακά στοιχεία τους για εγγύηση. Θα πρέπει να ε, αισθανόμαστε ε, συμπόνια για τους ανθρώπους αυτούς, για τους ανθρώπους. Μιλάμε για κλιματική αλλαγή, για κανόνες που τους επιβάλλουμε, μα εδώ τους έχει έρθει καταστροφή και συμφορά τους έχει βρει. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Σάιβερ. Χωρίς ήχο, δυστυχώς, η ομιλήτρια. vous parler, Madame Schreiber? Μπορείτε να πάρετε το λόγο, να μιλήσετε. Μιλάει ο μιλήτρια, αλλά δεν ακούγεται. We don't hear you. We can't hear you, Madame. Excuse me, Mrs. Schreiber, could you please try... Συγγνώμη, κυρία Schreiber. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί που λέει «Μιλήστε». Yes, I think it, it works now. Can you speak again? No, we can't hear you, madam. trying it's... Τώρα σας ακούμε, ναι. Τώρα δεν σας ακούμε. Ça πάρει, ça Μια τελευταία απόπειρα, αλλιώς θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες ε, στο μέλλον όταν θα ε, ε, ψηφίσουμε την έκθεση. Τελευταία απόπειρα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Well, uh, sorry for that. Looks like maybe... Συγγνώμη, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον εξοπλισμό που έχετε, ε, που έχουμε εμεί. Ευχαριστώ. Όπως σα είπα, αγαπητοί συνάδελφοι και εκπρόσωποι τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα έχουμε και άλλες ευκαιρίε να τα ξαναπούμε για το θέμα αυτό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τι αντίστοιχε πολιτικέ. Επίση, περιμένουμε έγκριση της διάσκεψης των Πρόεδρων για να γίνει μια κανονική έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και ο κύριος Μπόρκια, εισηγητής, θα μπορέσει να παρουσιάσει την θέση μας. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώνεται το τοπίο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στα πλαίσια του σχεδίου ανάκαμψης και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ακούμε και ακολουθούμε όλες τις στρατηγικές και τους στόχους, την πράσινη ανάπτυξη, την ψηφιοποίηση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικές ευκαιρίες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά χρειαζόμαστε στοχευμένες πολιτικές. Σας ευχαριστώ και πάλι αγαπητοί συνάδελφοι για τη σημερινή σας ε, παρουσία. Ήταν πολύ καλές οι συζητήσεις και πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που μας απασχόλησαν. Σας ευχαριστώ που σεβαστήκατε και το χρόνο σας, θαυμάσια. Και τελειώνουμε στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ, σας ε, αποχαιρετώ. Ε, μείνετε ασφαλείς, προσέχετε τον εαυτό σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά, την άλλη εβδομάδα, 4 Ιουνίου, στις 2 παρατέταρτο ώρα Βρυξελών. Γεια σας, όλα τα καλά.